κυβερνήτης ε, ε, Ουκρανικών αεροσκαφών που ήταν κρατούμενοι εδώ και αρκετό καιρό ε, απελευθερώθηκε σήμερα και η ερευνητική δημοσιογράφος η Καντίζα Ισμαήλοβα απελευθερώθηκε στο Αζερβαϊτζάν. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υπερασπιστεί με ιδιαίτερο στένος την απελευθέρωση αυτών των δύο θαραλέων γυναικών και επιτέλους μπορούμε να επιχαίρουμε διότι αυτές οι γυναίκες επιτέλους θα μπορέσουν να συναντηθούν με τις οικογένειές τους. Να συνεχίσουμε τις εργασίες. Πότε πότε έχουμε και καμιά καλή είδηση. Μας καθησυχάζει αυτό να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Τούν und Ευχαριστώ κύριε Κύριε Πρόεδρε.